δεν λειτουργεί Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που έχετε έρθει. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις στην ημέρησια διάταξη, θεωρώ ότι την έχουμε εγκρίνει, υπενθυμίζοντά σα ότι αύριο θα έχουμε μια πολύ σημαντική συνάντηση καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων για να συζητήσουμε τα θέματα της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ε, ασφάλειας μετά την ε, ισχύ της ε, συνθήκης Λισαβόνας και δει σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ των κοινοβουλίων. Ήδη είχα αναφέρει το θέμα αυτό τον Ιούνιο, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι ένας φάκελος πάνω στον οποίο πραγματικά πρέπει να ακουστεί η φωνή μας και σίγουρα και οι βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων που θα, ήρθαν, που θα έρθουν εδώ αύριο θα είναι σίγουρα εξαιρετικά ε, έτοιμοι και αποφασισμένα μας πούν ότι σε ό,τι αφορά την ΚΕΠΑ αυτοί είναι πλέον κατάλληλοι να έχουν ε, πιο ισχυρό λέγει από εμάς. Οπότε σας προειδοποιώ για να έχετε και εσείς τα αντίστοιχα επιχειρήματα αύριο να αντιτάξουμε. Θα, θα, δεχθούμε επίσης το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ γιατί έχουμε και ένα νέο σημείο ημερήσιας διάταξης που αφορά τη σχέση με το ΝΑΤΟ θα έχουμε και τον ειδικό εκπρόσωπο, τον επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Αφγανιστάν, τον ε, πρέσβη Ζατσκάς. Και για το, από το Συμβούλιο θα έχουμε τον Ολιβέο Σεστέλε, τον ε, Υπουργό Εξωτερικών για θέματα ευρωπαϊκά του Βελγίου και που όμως ε, θα είναι μέσω προσώπου, δεν θα μπορεί να είναι ο ίδιος μπροστά. Ευχαριστώ λοιπόν την προσοχή σα αύριο για την συνάντηση τη συνεδρία στην Αυριανή. Σήμερα ερχόμαστε στην ε, έκθεση που έχει προετοιμάσει η Κριστιαν Λέχ πάνω στην πολιτικοστρατιωτική συνεργασία και την ανάπτυξη πολιτικοστρατιωτικών ικανοτήτων. Μια πρώτη συζήτηση δυστυχώ εξαιρετικά βραχία και βεβαιασμένη έλαβε χώρα τον Μάιο και ζητώ συγγνώμη γιατί η Προεδρία μου δεν είχε καθόλου καλά οργανωθεί σε εκείνη την Ολομέλεια. Δεν είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να συζητήσουμε τον σημαντικό εκείνο φάκελο. Έχουμε όμως σήμερα την ευκαιρία και ζητώ από τον Κριστιαν να λάβει το λόγο για να μας ε, παρουσιάσει την έκθεσή του. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας παρουσιάσω σήμερα το προσχέδιο της ε, έκθεσης για την πολυκοστρατική συνεργασία και την ανάπτυξη πολιτικο-στρατιωτικών ικανοτήτων. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για τα πολύ κομπεντιμητικά σας σχόλια που έλαβα από πάρα πολλούς ε, ε, συναδέλφους. Προσπάθησα να κάνω τη διαδικασία αυτή στον πιο διαφανή. Οι σκιώδεις ηγητές έλαβαν νωρί την έκθεση αυτή, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση σήμερα. Και πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάρα πολλού εμπειρογνώμονε. Κάποιοι είναι εξ αυτών εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, το ΝΑΤΟ και από αρκετά κράτη-μέλη που είχαν την ε, ε, έβγαινε να μου, να μου παρουσιάσουν τις θέσεις των οργανισμών τους πάνω στο θέμα αυτό, την πολυξερωτική συνεργασία και πώς μπορούμε να κάνουμε δυνατόν πιο αποτελεσματική τη διεύθυνση διαχείρισης κρίσεων και σχεδιασμού. Έχω την εντύπωση ότι όλοι οι συνομιλητές θέλαν πάρα πολύ να συνεισφέρουν στην έκθεση αυτή, γιατί είναι ιδιαίτερη σημασία στο θέμα αυτό, ιδιαίτερη εν ώψη των διαπραγματεύσεων για την μελλοντική δομή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης η πολιτικοθεωρητική συνεργασία είναι πολύ ευρύ όρο και μπορεί κανεί να φανταστεί πάρα πολλά πράγματα υπό τον όρο αυτό. Θα ήταν ανόητο να προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε όλα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να εστιάσω την έκθεση αυτή πάνω σε πολύ συγκεκριμένα απτά θέματα. Καταρχά, ό,τι αφορά τον, τον θεσμικό συντονισμό των εφιστάμενων ευρωπαϊκών εργαλείων. Δεύτερον, στην ανάπτυξη πολιτικοθεωρητικών ε, ικανοτήτων για τη διαχείριση κρίσεων και τρίτον στη διασφάλιση του ότι θα υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα για τη ε, ε, διαχείριση κρίσεων, πολιτικοθεωρητικών κρίσεων. Η έκθεση μου λοιπόν είναι δομημένη σύμφωνα με αυτά τα τρία πεδία. Μπορεί βέβαια κάλλιστα να σκεφτούμε και πάρα πολλά θέματα σε ό,τι αφορά το πλαίσιο πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας, όπως των σχέσεων μεταξύ στρατιωτικών δυνάμεων και μη κυβερνητικών οργανισμών, αλλά είναι τελείως διαφορετική η διάσταση του θέματος αυτού. Νομίζω ότι η έκθεση θα έχανε από την στόχευσή τη εάν προσπαθούσαμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα από κοινού. Οι περισσότεροι θα συμφωνήσουμε βέβαια ότι, η, ότι στην ΚΕΠΑ ε, απαιτείται πολύ καλύτερος και είναι επιθυμητός ως καλύτερος συντονισμός των, στα θέματα πολιτικοστατικής συνεργασίας. Στις πρώτες παραγράφους ε, μέχρι το 2014, κοιτάω τους τρόπους του πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί στην θέσπιση ακριβώς της ε, ε, υπηρεσίας, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω εδώ. Οι σχετικές ανισορροπίες που πιστεύω υπάρχουν στις διάφορες δομές. Καταρχάς, πολύ μεγάλη πλειοψηφία ε, αποστολών ε, επιτελείων σχεδιασμών είναι μάλλον πολιτική υφή και αυτό δεν εκατοπρίζεται επαρκώ στι δομέ η Διεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Σχεδιασμού, μάλλον συγγνώμη, το Επιτελείο Σχεδιασμού και Εκτέλεση των Πολιτικών Δράσεων έχει μόνο 60 άτομα. Η στρατιωτική πτυχή δεν έχει καθόλου εμπειρογνώμονες πάλι σε όλες τις προτεραιότητες που τίθεται σε ό,τι αφορά τις πολιτικές δράσεις, όπως είναι η αστυνομία, η δικαιοσύνη και την πολιτική διοίκηση. Προσθέτως φαίνεται ότι η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ του στρατηγικού σκέλους και του επιχειρησιακού σκέλους φαίνεται να είναι ασαφής και γι' αυτό ζητώ καλύτερο καθορισμένη στρατηγική. Και, γι αυτό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτή τη στιγμή τα κοινοβούλια είναι υπεύθυνα και αρμόδια να συμμετάσχουν στη συζήτηση αυτή. Κατά δεύτερο πιστεύω ότι θέλουμε να είμαστε σοβαροί σε ό,τι αφορά την πολιτικοστρατιωτική συνεργασία. Πρέπει σίγουρα να έχουμε μια μόνιμη δομή επιχειρησιακού σχεδιασμού και διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι το Κοινοβούλιο αυτό ζητά να υπάρξει ένα κεντρικό ε, στρατηγείο για μια αποστολή επιτήρησης δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να συνδέεται πάρα πολύ στενά στην ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και ίσως κάποιο είδους αν θέλετε διεύθυνση διαχείριση κρίσεων και σχεδιασμού. Ταυτόχρονα όμως είναι ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι οι ιδιαιτερότητες κάθε τομέα και κάθε ειδικότητα θα γίνονται σεβαστές και να μην ε, υποτάσσουμε το πολιτικό προσωπικό στο στρατιωτικό σχεδιασμό ή αντιστρόφω. Στο δεύτερο κομμάτι της εκθεσης παραγράφου παραγράφους 15-31, εστιάζω στην ανάπτυξη πολιτικών και στρατιωτικών ικανοτήτων. Νομίζω ότι υπάρχει σαφής, ε, σαφές κενό μεταξύ αυτών τα οποία δεσμεύτηκαν να παράσχουν τα κράτη-μέλη και αυτών που πραγματικά έχουν διαθέσει στις ευρωπαϊκές αποστολές. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία στο κενό αυτό γιατί μπορεί να αποτελέσει ένα μελλοντικό πολιτικό πρόβλημα και πρακτικά δεν έχουμε τα μέσα να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τους ε, στόχους που έχουν τεθεί. Για παράδειγμα, τα κράτη-μέλη ήδη το 2004 ε, δεσμεύτηκαν να κάνουν και να διαθέσουν πάνω από 11.000 ε, πολιτικό προσωπικό. Όμως είναι πασίγνωστο ότι ακόμα και οι υφιστάμενες πολιτικές αποστολές που, απο, απασχολούν περίπου 3.000 άτομα τη στιγμή, υποφέρουν από διαρκή έλλειψη προσωπικού εκατοντάδων ατόμων. Ω εκ τούτου γίνεται έκκληση στην έκθεση αυτή στα κράτη-μέλη να αντισταθμίσουν την κατάσταση αυτή και να μην θέσουν άλλου πιο φιλόδοξου στόχου προτού διασφαλίσουν ότι πραγματικά θα εκπληρούν τι ε, δεσμεύσει που έχουν αναλάβει. Διαφορετικά, οι στόχοι δεν θα είναι αξιόπιστοι. Και αυτό σημαίνει ότι εν γέννη η ευρωπαϊκή πολιτική δεν είναι αξιόπιστη το πολιτικό προσωπικό που συμμετέχει σε τέτοιε αποστολέ είναι σε θελοντική βάση. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλουμε περισσότερου αστυνομικού και δικαστικού διαθέσιμου για τι αποστολέ αυτέ, τα κράτη-μέλη θα πρέπει καταρχά να εξασφαλίσουν ότι η εμπειρία την οποία θα αποκομίσουν θα γίνεται σεβαστή και θα εκτιμάται. Αυτό σημαίνει όχι μόνο στα θέματα των αμοιβών, αλλά και στι προοπτικέ μελλοντική του αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο και όλα τα αρμόδια, τα συναρμόδια υπουργεία θα πρέπει να συνεργαστούν για να ε, έχουν σχετικές στρατηγικές για το μέλλον. Κάτι άλλο θεμελιώδες είναι η εκπαίδευση. Και υπάρχουν καλά παραδείγματα από διάφορα κράτη-μέλη που τονίζονται στην έκθεση, το βλέπουμε στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν μπορώ να διατρέξω τώρα όλα τα σημεία. Θα ήθελα λοιπόν μόνο να τονίσω δύο ακόμα θέματα από αυτήν την άποψη. Πρώτον, είναι η όλη έννοια ε, ενοποιημένων ε, αστυνομικών ε, μονάδων που είναι πολύ κέρυες στην όλη συζήτηση για το συνδυασμό πολιτικών και στρατιωτικών μέσων στην διαχείριση κρίσεων. Αυτές οι μονάδες μπορούν να είναι πάρα πολύ ευέλικτες και μπορούν ίσως να τεθούν και υποστρατιωτική στρατιωτική διοίκηση. Οπότε είναι μια έννοια που φαίνεται να είναι η πλέον κατάλληλη για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα ε, κατεπηγουσών καταστάσεων. Και πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να προάγω την, ε, την, ε, γερμανικό, ε, γερμανι, την ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων με πολιτικές δυνάμεις όπως είναι ε, στη Διεθνή Ειρηνευτική Δράση που συνδυάζεται το από το Γερμανικό Κέντρο Αστυνομίας και Χωροφυλικής. Ένα δεύτερο σημείο είναι η Ευρωπαϊκή Δύναμη Χωροφυλακής και ένα δεύτερο είναι οι ομάδες κρούσης. Οι πολιτικές ομάδες αντίδρασης της κρίσης. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη ε, χρηματοδότηση βέβαια για να γίνεται καλύτερη χρήση των μονάδων αυτών. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν πάνω σε κοινή χρηματοδότηση κάθε δαπάνη τέτοιων ε, αποστολών, τέτοιων διαδικασιών. Διαφορετικά η συμφωνία για την, ε, για την ε, δρομολόγηση τέτοιας αποστολής δεν θα μπορεί να γίνει ποτέ, γιατί τελικά κανείς δεν θα θέλει να καλύψει τα διδαπάνες. Αυτές λοιπόν οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να μετασχηματιστούν σε μακρόπνοες συνεργασίες, όπως αντίστοιχα όπως έγινε πριν με τις, ε, με τις δυνάμεις της, ε, των ε, σκανδιναβικών χωρών, όπως είχε γίνει στο παρελθόν. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν επίσης οι ομάδες αυτές σε ενδεχόμενες ε, δράσεις κατεπηγόντων και αντιμετώπισης ε, καταστροφών και βέβαια σε ευθυγράμμιση με τις ε, γραμμές του, της Συμφωνίας του Όσλο. Τώρα, στο τρίτο κομμάτι που είναι για μια ευρεία αντιμετώπιση των κρίσεων, αντιμετωπίζονται θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Προφανώς θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η στενή συνεργασία ε, για πολιτικέ και ιδιωτικέ επιχειρήσεις, αλλά μόνο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη δυνατοτήτων διαχείριση κρίσεων. Τονίζω ότι για άλλη μια φορά μπορούν να επιτευχθούν και να εκμεταλλευτούμε πάρα πολλέ ε, συνέργειες μεταξύ των ε, διαφόρων κομματιών έρευνα και τεχνολογία στο πολιτικό και στο ερωτικό σκέλος. Αλλά θα πρέπει να, να θυμόμαστε πάντα ότι υπάρχουν περιορισμένοι πόροι σε ό,τι αφορά τα ερευνητικά προγράμματα έρευνα και τεχνολογία στα θέματα ε, άμυνας θα πρέπει να φανηθεί συνεργασία ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση ε, διαστημικών ικανοτήτων, τα μη επανδρομένα χήματα και την ε, διαθαλάσσης ε, επιτήρηση. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει η διάθεση εξοπλισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να είναι άμεσα διαθέσιμα Στου εξοπλισμούς όταν χρειαστεί, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για πολιτική ή στρατιωτική αποστολή. Κάποιος εξοπλισμός όμως ίσως πάρα πολύ γρήγορα να απαρχαιώνεται. Επομένως η απόφαση θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται επί τη βάση μιας ανάλυσης κόστους ωφέλης για κάθε είδους εξοπλισμό. Γι' αυτό ζητώ να υπάρχουν τέτοιου είδους αναλύσεις οι οποίες θα πρεπει παντα να λαμβανεται επι τη βαση μιας αναλυσης κοστους ωφελης για καθε ειδους εξοπλισμο γι αυτο ζητω να υπαρχουν τετοιου ειδου αναλυσεις οι οποιες θα καθοριζουν για τι είδους ε, εξοπλισμού ποια αποθήκη είναι η βέλτιστη και ίσως κάποιες άλλες λύσεις όπως συμφωνίες πλαίσιο με προμηθευτές ή ε, μήπως ε, εξοπλισμός που θα δίνεται ad hoc από συγκεκριμένα κράτη-μέλη ανάλογα με τις ε, ε, καταστάσεις. Είναι και... Είχαμε μια μέση, στην μέση εξέταση, στην ενδιάμεση εκθέση του, του προϋπολογισμού, μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε. Έχω ολοκληρώσει την έκθεση, την αφιερωμένη στι δύο πιο συγκεκριμένε εταιρικέ σχέσει με, με τον ΟΗΕ και τον ΝΑΤΟ. Θέλω να τονίσω ένα τελευταίο σημείο εδώ. Του κατά πόσον θέλουμε ή, ο, θέλουμε είτε όχι, το ΝΑΤΟ ε, σκέφτεται επίσης να επισέλθει στο πεδίο της διαχείρισης πολιτικών κρίσεων. Ο μεγαλύτερος ελιγμός ε, πολιτικής κρίσης και διαχείρισης κρίσης ε, του ΝΑΤΟ έλαβε χώρα στην αρχή του έτους. Και μία από τις εικασίες, αν θέλετε, τα επιχειρήματα του ΝΑΤΟ είναι ότι είναι ανύπαρκτη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του σημερινού κόσμου. Αυτό που θεωρώ ότι θα ήταν πολύ μεγάλο λάθο θα ήταν να αφήσουμε τον ΝΑΤΟ να αρχίσει τι δικέ του διαδικασίε, αμυγό δικέ του σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων για διαχείριση πολιτικών κρίσεων που θα οδηγούσε σε πάρα πολλέ επικαλύψει και διπλασιασμό προσπαθειών. Γι' αυτό λέω στην έκθεση ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να μπορεί να βασίζεται στι ικανότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποια πεδία. Η μορφή της ε, υποστήριξης αυτή μένει να ιδωθεί και να διαπομορφωθεί, αλλά θα πρέπει να είναι κομμάτι της συνολικής ε, συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Ο στόχος όλων αυτών είναι καλύτερος συντονισμός ε, πολιτικών και στρατιωτικών μέσων ε, στα πλαίσια της ΚΕΠΑ. Νομίζω ότι μπορεί να είναι πολλά πράγματα αντιφατικά, αλλά νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να τα αποκρίνεται στην κράση με επαρκή εργαλεία, με επαρκή μέσα και να μπορεί να τα αποκριθεί ε, συνεκτικά. Αυτή τη στιγμή, στο... εάν υπάρξει IT δεύτερου τύπου στον ΟΗΕ τέτοιας διάστασης και τόσο προβληματική και οι Αμερικανοί δήλωναν μέσα στον ΟΗΕ ότι η διασπορά των ικανοτήτων, των, των δυνατοτήτων τους δεν είναι ικανοί, δεν είναι επαρκείς και επομένω χρειάζονται τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωση. τελικά εμείς δεν θα μπορούσαμε να αποκριθούμε και να αναλάβουμε το ρόλο αυτό. Η δημιουργία λοιπόν μιας ε, τέτοιας ΕΕΔ ε είναι σημαντική. Η ανάπτυξη ε, τέτοιων δυνατοτήτων είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σημαντικό κομμάτι ε, που θα ενισχύσει την ΚΕΠΑ. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπληρώσει τους ε, στόχους αυτούς προτού θέλει να εισάγει νέους και πιο φιλόδοξους. Περιμένω και ευχαρίστω τα σχόλιά σας και θα ήθελα να υπάρξει μεγάλη συνένεση στο θέμα αυτό γιατί υπό την παρούσα κατάσταση όπου μπορούν πραγματικά να αποφασίσουμε επί σημαντικών θεμάτων δίνει σημαντική ισχύ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστούμε πολύ, Κριστιαν Έλλερ. Νομίζω ότι πράγματι είναι μια πολύ σημαντική έκθεση που φύγει σημεία επί των οποίων εξάλλου υπάρχει μεγάλη συνένεση ως προς την ουσία του θέματος. Ε, οι περισσότερες ομάδες, το σύνολο των ομάδων, ήθελα να συνταχθεί μια τέτοια έκθεση, διότι είναι πολύ σημαντική διότι μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχουν μάλλον διατάξεις στη συνθήκη που επιβάλλουν αυτόν τον συντονισμό πολιτικού στρατιωτικού χαρακτήρα και θα πρέπει το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας να αποφανθεί επί αυτών των σημείων. Με αρκετοί συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Δίνω το λόγο στον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Μαυρονικόλα, που ήταν και σκιώδης από πλευρά σοσιαλιστών. Απλώς χωρίς να επαναλάβουμε όλα τα σημεία του κειμένου, να πούμε καταρχήν ότι ο φίλος ο Κρίστιαν πράγματι ανταποκρίθηκε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό για ένα θέμα το οποίο είναι άκρος νεοφανές στην Επιτροπή μας ότι υπήρξε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων αλλά πολύ περισσότερο ότι και το ίδιο το κείμενο είναι δομημένο με τρόπο ικανοποιητικό αγγίζοντας όλα εκείνα τα σημεία τα οποία χρειαζόταν και πολύ περισσότερο αναφερόμαστε σε, μια, σε ένα ρεπορτ, το οποίο αναφέρεται για πρώτη φορά σε μια πολιτικοστρατιωτική συνεργασία. Το θέμα είναι καινούριο και νομίζω ότι αυτό το κείμενο στους βασικούς του παράμετρους αντιπροσωπεύει την κοινή αντίληψη. Θα υποσημείωνα ότι πράγματι υπάρχει ανάγκη για να υπάρχει μία μόνιμη δομή, μία, ε, να υπάρχουν εγκαταστάσεις τέτοιες οι οποίες να δίνουν την δυνατότητα ταχείας ενεργοποίησης και πραγματικά εντός του κειμένου αυτού αναφέρονται οι αδυναμίες οι οποίες υπάρχουν. Ένα δεύτερο σημείο έχει σχέση να κάνει με την τεχνολογία και πολύ περισσότερο με την ανάγκη χρηματοδότησης αυτών των επιχειρήσεων και ένα τρίτο μέρος αναφέρεται στην ε, πραγματική δυνατότητα που πρέπει να υπάρξει η αδιάθεση κοντινίων και καλύτερη συνεργασία με μεγάλους παγκόσμιους οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη και τον ΝΑΤΟ οι παρατηρήσεις από τη σοσιαλιστική ομάδα είναι επιμέρους. Ε, θα συγχαρώ και εγώ τον ε, Χριστιαν για την παρουσίαση αυτού του κειμένου και νομίζω ότι το κείμενο αυτό αποτελεί την βάση για να ξεκινήσουμε ε, και να αντιμετωπίσουμε ορθά το θέμα των, της πολιτικοστρατιωτικής δράσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε. Η κυρία Νέιτς. Ο κύριος Βαμπάλεν ήταν ο Σκιώδης, αλλά δεν είναι σήμερα εδώ. Νομίζω ότι συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις στη Χάγη, αν δεν κάνω λάθος. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή τον κύριο Έλερ για την εξαιρετική αυτή η έκθεση που αποτελεί ένα κρίκο στην εξέλιξη των ιδεών μας και των θέσεών μας σε σχέση με την συνεργασία ως προς το στρατιωτικό και πολιτικό σκέλος για θέματα κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Εδώ και αρκετό χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι υπάρχει επαρκή συνέργεια στο στρατιωτικό και πολιτικό τομέα. Θα ήθελα να αναφερθώ στη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που παρουσίασε την κατάσταση σε μια συνεδρίαση η οποία παρεξετράπει κάπως, αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση την προηγούμενη εβδομάδα, όπου αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει, και αυτό το λέω εγώ, μια πολιτική, μια δυνατή πολιτική άμυνας και ασφάλειας στη δική του θέση, θα μιλούσα για την κατάρτιση μιας πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, η οποία αρχίζει να παίρνει μορφή. Δεν ε, έχει διατρανωθεί. Εν πάση περιπτώσει αυτό το θέμα είναι σημαντικό διότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στις εξελίξεις και ο συνάδελφος τονίζει ότι τα κράτη-μέλη ε, παλινοδούν και καθυστερούν ως προς την επίτευξη των στόχων που όμως είχαν εγκρίνει σε σχέση με το σκέλος των πολιτικών ικανοτήτων. Και αυτό ίσως μας εκπλήσει, αλλά είναι και κατανοητό σε τελευταία ανάλυση, διότι είναι ε, δύσκολο να υπάρχει μία εξωτερική αποστολή εκτός ε, επικρατείας Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρατιωτικών, δικαστικών, αστυνομικών ε, αρχών ή άλλων δυνάμεων του πολιτικού σκέλους. Αυτό είναι κατανοητό, γιατί για μια χώρα ε, όπου επικρατεί η ειρήνη, οι στρατιωτικοί βρίσκονται στους στρατώνες, δεν χρειάζεται να μεταβούν κάπου αλλού. Και οι δικαστικές αρχές και οι αστυνομικές λειτουργούν καλώς. Κάπως εξεπλάγιν όταν διάβασα αυτή την έκθεση και όταν άκουσα τον συνάδελφο που μας είπε ότι ως προς το ε, στρατιωτικό σκέλος. Η λέξη battle group δεν υπάρχει πια. Με βάση την προηγούμενη θητεία και ο προκάτοχός σας, ο κύριος Ντανζόν, μας ε, είχε πει πολλά και σημαντικά και είδα ότι αυτός ο όρος δεν υφίσταται πλέον. Και du volet militaire, c'est une des questions sur il faudrait quand même que nous nous... Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ισχύει πια αυτός ο, ο όρος για τις σκανδιναβικές χώρες, δηλαδή για τα Nordic Battle Groups. Ποια είναι τα εμπόδια ε, που δεν συντελούν στο να χρησιμοποιούνται. Γιατί οι αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων ίσως αντιμετωπίσουν δυσκολίες να ε, προβούν στη σύσταση ενός στρατιωτικού σκέλους από που να παρτίζεται από εθνικές ένοπλες δυνάμεις. Αλλά είναι πολύ κρίμα να έχουν συσταθεί αυτές οι ομάδες και μετά ε, να μην χρησιμοποιούνται αυτές οι μάχημες ομάδες. Θα ήθελα να σταθώ και στο θέμα της Eurocore, που ξέρω ότι βρίσκεται εκτός αυτού του πλαισίου. Υπάρχει όμως αυτή η δομή εκτός Στρασβούργου που έχει καινούριο υλικό, διαθέτει καινούριο υλικό το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Και είναι πολύ κρίμα γιατί υπάρχουν ε, πολλά ερωτηματικά που θα πρέπει να μας αποσχολήσουν. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να προβεί σε έναν απολογισμό. Ίσως εμείς να μην είμαστε στη σωστή θέση διότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε προκατηλημένοι, δεν είμαστε προειδεασμένοι. Αλλά στην αρχή είχαμε τις 60.000, ε, την καταλείπουμε αυτή την σειρά, μετά τα battle groups τα εγκαταλείπουμε και τώρα βρισκόμαστε σε μια τρίτη γραμμή. Τι κάνουμε. Θα πρέπει λοιπόν να εμβαθύνουμε το όλο ζήτημα έτσι ώστε να μην λέμε ότι διαθέτουμε στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίες είναι μάχημες, αλλά έμπρακτα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτά είναι τα πρώτα σχόλια που θα ήθελα να αναφέρω. Ο συνάδελφος έχει απόλυτα δίκιο όταν λέει ότι στα πλαίσια των σχέσεων ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης το ΝΑΤΟ θα προσπαθήσει να προβεί σε σύσταση ενός πολιτικού σκέλους. Δεν είναι πρωταρχικό του έργο και δεν βρίσκεται στη σωστή θέση για να επιτύχει κάτι τέτοιο. Αυτό δεν θα ήταν δυνατόν, δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό. Πολλοί συνάδελφοι που συμμετέχουν στις συνελεύσεις ΝΑΤΟ ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουν ότι υπάρχει ένα είδος ανταγωνισμού μεταξύ των δύο. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Έλλερ και επειδή δεν υπάρχουν ούτε προειδεσμοί ούτε ιδεολειψίες, θα πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω το θέμα. Γιατί δεν έγινε χρήση των battle groups, των μάχημων ομάδων. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ε, λόγος γι' αυτό. Γιατί ζητάμε από τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους ως προς τη διάθεση προσωπικού, αστυνομικού, ε, δικαστικών και άλλων ε, προσώπων που να εκπροσωπούν το πολιτικό σκέλος και όχι το στρατιωτικό και από την άλλη υπάρχει μία κλιμάκωση και πώς μπορούμε να μεταπίσουμε το ΝΑΤΟ έτσι ώστε να μην ακολουθήσει το πολιτικό σκέλος. Κάτι το οποίο δεν καταφέρουμε. Ό,τι ισχύει για τους στρατιωτικούς ισχύει και για τους δικαστικούς. Δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν δηλαδή δικαστικοί που διαθέτουμε στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους που θα υπηρετούν το ΝΑΤΟ, άλλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι το ΝΑΤΟ. Το ίδιο ισχύει και για το στρατιωτικό σκέλος. Θα πρέπει λοιπόν να εξεύρουμε έναν τρόπο έτσι ώστε να αποσαφινιστεί η κατάσταση και όσον αφορά το Eurocore. Ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα σχόλια σε σχέση με το Eurocore, νομίζω ότι γνωρίζετε ότι στην επόμενη Ολομέλεια στο Στρασβούργο θα έχουμε την δυνατότητα να μεταβούμε την Πέμπτη το απόγευμα και θα ήθελα να αλλάξουμε κάπως τα ωράρια έτσι ώστε να μπορέσουμε να, ψηφούμε, να ψηφίσουμε και μετά να μεταβούμε στη Eurocore, στην έδρα της Eurocore που δεν χρησιμοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθεί στους συμπολίτε μας. Κυρία Λέζιν, έχει το λόγο. Ja, vielen Dank. Ähm, Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς πρέπει ευθύ εξ αρχής να αποσαφηνίσω και να πω ότι η δική μου κοινοβουλευτική ομάδα, η Ενωτική Αριστερά, και εγώ η ίδια, αυτή την έκθεση με κανένα τρόπο δεν θα μπορέσουμε να την εγκρίνουμε υπάρχει ουσιαστικά δεν υπάρχει ούτε ένα και μόνο σημείο σε αυτή την έκθεση που να μην είχαμε ενστάσεις και αντιρρήσεις. Και έτσι με τροπολογίες θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε τα πράγματα. Θα ήθελα σύντομα να αναφερθώ στα μεγαλύτερα σημεία επικρίσεων που έχουμε να διατυπώσουμε. Στο άρθρο 8 και το άρθρο 29 πρώτα απ' όλα με το αίτημα της διεύρυνσης ε, σε σχέση με την στρατιωτική ανθρωπιστική βοήθεια και την ε, συνδρομή, άμεση συνδρομή. Το ότι η ΑΕΤ ακριβώς βρίσκεται εδώ, σε αυτό το πλαίσιο ως υπόδειγμα, ως παράδειγμα, δείχνει σαφέστατα ότι δεν έχουμε πείρα με τις πρακτικές ε, και με το τι γινόταν στο παρελθόν και έχω καμιά φορά την εντύπωση ότι δεν μπορεί κανείς με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσει πείρα ή ότι δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ε, ε, βασιζόμαστε και να οικοδομούμε. Για την IT ε, πρόκειται λοιπόν για μια εσφαλμένη ερμηνεία των συμβάντων. Έχουμε πολυάριθμες εκθέσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων που λένε ότι οι στρατιωτικοί δεν ήταν αναγκαίοι να είναι παρόντες. Και μάλιστα με την παρουσία τους οδηγήθηκαν στο να κλείσει το αεροδρόμιο και να μην μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Σας ερωτώ λοιπόν τώρα, πώς μπορεί αυτή η επίκριση, αυτές οι κριτικές, πώς μπορούν να συμβιβαστούν με τα αιτήματά σας, με τα πρακτικά αυτά βιώματα τα οποία είχαμε στο παρελθόν. Πώς μπορούν όλα αυτά να ενταχθούν σε αυτή την έκθεση με αυτόν τον τρόπο. Η δεύτερη επίκριση αφορά το αίτημα για ένα λειτουργικό γενικό επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 12 και η σύμπτυξη των πολιτικών και στρατιωτικών δράσεων όσον αφορά τον προγραμματισμό, για παράδειγμα στο άρθρο 13. Ιδιαίτερα προβληματικό είναι το ότι στο άρθρο 13 προτείνεται ένα γενικό επιτελείο να δημιουργηθεί για την διαχείριση κρίσεων. Και εδώ πρόκειται για τις λειτουργικές ε, δυνατότητες σχεδιασμού στρατιωτικών αποστολών αλλά και πολιτικών αποστολών. Αλλά επίσης και την συγχώνευση, για την κάλυψη του τομέα της ασφάλειας ε, και σε σχέση με το Planning Directorate, δηλαδή το ε, ε, επιτελείο σχεδιασμού δράσεων που θα δράμε με αυτόν τον τρόπο. Ναι, μεν τονίζει το άρθρο 14 ότι υπάρχουν διαφορετικές αλυσίδες εντολών που διασφαλίζονται στην ιεραρχία εντολών και ότι θα έχουμε μια ένα πολιτικό σκέλος και ένα στρατιωτικό σκέλος που θα λειτουργούσαν. Όμως παρόλα αυτά δημιουργείται ένα βήμα συγχώνευσης πολιτικής και στρατιωτικής διαχείρισης Συγχωνεύονται αυτά, πράγμα το οποίο εμείς απορρίπτουμε. Αυτή η συγχώνευση ή αυτός ο συμφυρμός είναι κάτι το οποίο εμείς είχαμε προειδοποιήσει ότι δεν έπρεπε να γίνει. Και σήμερα το τελευταίο σημείο επίκρισης αφορά το άρθρο 30, Την διεύρυνση δηλαδή μέχρι την απόλυτη κάλυψη των ε, δαπανών και των ε, εξόδων. Μια και μέχρι σήμερα ένα μικρό μονομέρος του κόστους στρατιωτικών ή πολιτικών στρατιωτικών δράσεων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μέσω του μηχανισμού Ατένα-Αθηνά καλύπτονται οι μεγάλες ε, χώρες που διαθέτουν ε, ε, ενόπλους ενδιαφέρονται να υπάρχει η κατανομή, ο επιμερισμός των δαπανών. Η δική μας κοινοβουλευτική ομάδα είναι εναντίον του να διευρυνθεί ο επιμερισμός δαπανών μέσω της δυνατότητας Αθηνάς. αυτά είναι, ας το πω έτσι, τα κυριότερα σημεία κριτικής που έχουμε να διατυπώσουμε και στη συνέχεια αυτά θα γίνουν πιο σαφή με τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ε, παρουσιάσατε την κριτική σας, την γνωστή, αν μου επιτρέπετε να πω, γιατί είχατε ήδη την ευκαιρία να επαναλάβετε τα σχόλια αυτά κατά επανάληψη. Προβληματίζομαι λίγο από την κριτική σας σε ό,τι αφορά την ΑΕΤ. Γιατί εάν είχε χρησιμοποιηθεί στρατιωτικός εξοπλισμός στην ΑΕΤ, δεν είχε χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς λόγους. Οι στρατιωτικοί δηλαδή οι οποίοι λειτουργήσαν στο αεροδρόμιο ή στην ανοιχτά της θάλασσας της ΑΕΤΗΣ δεν έγινε για τους ίδιους στρατιωτικούς λόγους, αλλά για να φέρουν επιστημιστική βοήθεια και να βοηθήσουν στην ε, φοδιαστική αλυσίδα. Και αμφιβάλλω κατά πόσο οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί που αναφέρατε εσείς είχαν τα εναέρια ή θαλάσσια μέσα για να μπορούν να αναλάβουν τόσο βαγγές αποστολές. Προβληματίζομαι λίγο. Αντίθετα, πιστεύω ότι η ΑΕΤ καταδεικνύει το των αναγκών που απαιτούνται σε τέτοιου είδου κρίσει, για να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδου κρίσει και θα μπορούσαμε που να μην χρησιμοποιήσουμε στερεωτικά μέσα. Το κατά πόσο τα ελικόπτερα είναι στερεωτικά ή όχι, ομολογώ ότι εφόσον σώζουν ζωέ, ζωέ δεν με ενδιαφέρει ποσό. Όπω το είδαμε και με το σεισμό στο Πακιστάν με τον ΝΑΤΟ, όπω το είδαμε στι πλημμύρε ομολογώ ότι λίγο προβληματίζομαι από την χρήση του παραδείγματος αυτού που κάνετε, που κατ' εμέ αντιθέτως διατρανώνει ακριβώς την πολύ μεγάλη ανάγκη που υπάρχει συνεργασία στρατιωτικών και πολιτικών μέσων. Ούτως ή άλλως, αν πρόκειται για στρατιωτικά μέσα, δεν είναι για στρατιωτικές δραστηριότητες, αλλά χρησιμοποιούνται προς όφελος και για τη διοργάνωση ε, πρώτων βοηθειών και για επιστημιστική βοήθεια. Ενδεχομένω να κάνω λάθος. Τι να πω, αλλά έτσι νομίζω. Ο Γκάλερ, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. σε αυτό το είχα σκεφτεί ότι ο συνάδελφος Έλερ τις επικρίσεις της συναδέλφου θα τις είχε εκ προημίου αντιμετωπίσει λάβει υπόψη αν λέγαμε ότι δημιουργήθηκε, σε δημιουργήθηκε στενοπός στο αεροδρόμιο λόγω της παρουσίας στρατιωτικών εδώ έχει αναφερθεί improved coordination, ε, βελτιωμένο συντονισμό σε σχέση με τη δράση στην ε, IT. Ίσως έτσι με αυτόν τον τρόπο από τα lessons learned, τα συμπεράσματα που έχουμε συναγάγει, θα μπορούσαμε να είμαστε πιο, ας το πω έτσι, σωστοί. Αλλά ως θέμα αρχής δεν θα εκπλαγείτε ότι ο συντονιστής του ΕΛΚ την έκθεση του συναδέφου μου εδώ την θεωρώ πολύ θετική και την ε, υπερψηφίζω. Και όπως και αναφέρθηκε και στους περισσότερους συναδέλφους προηγούμενα, όλα αυτά τα σημεία και όλα τα θέματα τα οποία αναφέρονται όσον αφορά ελλείψεις ή ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν είναι ανάγκη να καλυφθούν, πρέπει να γίνουν αυτές οι δράσεις και για το Nordic Battle Group το οποίο αναφέρθηκε πιο πριν θυμάμαι υπό την ε, Σουηδική Προεδρία που είπε ο Καρλ Μπίλτζ ότι θέλω να δω ότι θα υπάρξουν και ότι θα δημιουργηθούν και θα λειτουργούν αυτές οι μονάδες. Και μπορούμε να φανταστούμε για το, για το ότι αυτή η αρχή για την δημιουργία, το ποιο, ποιος θα είναι αρμόδιος για τη συμμετοχή σε αυτά τα battle groups, για εκείνους που θα συμμετέχουν όταν έρχεται η σειρά τους, ε, δεν είναι η πιο ευχάριστη κατάσταση. Καμιά φορά ε, και για την δράση, για παράδειγμα στο Κονγκό, όταν θα ήταν η σειρά της Γερμανίας ε, να αποστείλει τέτοιες δυνάμεις ή να διαθέσει τέτοιες δυνάμεις, ε, πώς να το πω, αποφασίστηκε, ελήφθη απόφαση υπέρ ενός άλλου προτύπου, ενός άλλου μοντέλου θα έπρεπε να σκεφτούμε για τις δομές αυτές τις οποίες θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και στο τέλος. Use them or lose them, δηλαδή γιατί διαφορετικά χάνεται η δυνατότητα αν δεν χρησιμοποιηθεί η, δυνατο... η... η παρουσία αυτών των μονάδων. Τώρα και για την ε, παρουσία αυτών των ε, ε, δυνάμεων και εδρών και στο στετίν είναι διαθέσιμες για πιθανές τέτοιες δράσεις αλλά μέχρι στιγμής από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν κληθεί να δράσουν. Και μέσα στο πλαίσιο ενός, ας το πω έτσι, πλαισίου αμυντικών δράσεων, ο υπεύθυνο του Eurocore, του Ευρωσώματος στο Στρασβούργο, βρίσκεται καθοδόν και αποσαφηνίζει με τον πιο κατάλληλο ενδεδειγμένο τρόπο ότι υπάρχει εκεί ένα δυναμικό στο Στρασβούργο και ότι η δική μας δουλειά είναι να συναγάγουμε τα συμπεράσματα και πολιτικά, πολιτικά να ε, συναγάγουμε τις ε, ευθύνες μας, να συνάξουμε τις ευθύνες μας, να δούμε με ποιο τρόπο θα πρέπει να δράσουμε, να κινητοποιηθούμε αν χρειαστεί. Κατά τούτο θα έλεγα ότι η κρίση ε, ο σχεδιασμός πολιτικών δράσεων και πολιτικών δράσεων στη νέα δομή συμπτύσσονται ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός από την ΕΕ στρατιωτικά και πολιτικά συνδυάζεται. Αλλά για την εκτέλεση δράσεων έχουμε τα εθνικά επιτελεία στα οποία προσφεύγουμε. Και θα πρέπει να δούμε εδώ και με το, την δράση Αταλάντη και στο συνδυασμό ΕΕ και ΝΑΤΟ πώς μπορούν να, αποκτήσουν σάρκα και οστά και να δράσουν. Και θα ήταν καλύτερο θα έλεγα αν όλα υπό ένα πρίσμα και με μία, ας το πω έτσι, με ένα μοντέλο, με ένα πρότυπο μπορούσαμε να τα ε, καλύψουμε ως δράσεις. Με ένα ενιαίο πρότυπο. Κατά τα άλλα, μία ερώτηση θα είχα. Ίσως μία πρόταση ως ερέθισμα να δώσω μέσα στο πλαίσιο της ε, πληρέστερης ολοκλήρωση ε, εκείνων που έχουμε υπό τις συνθήκες Λισαβόνας. Μία αναφορά ίσως ε, της European Defense Agency να γίνει στο κείμενο σε κάποιο σημείο. Είναι ένα σημαντικό μέσο, ένα σημαντικό εργαλείο μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της συνθήκης Λισαβόνας. Και η ρήτρα συνδρομής ε, είναι και αυτό σημαντικό στοιχείο να ε, αναφέρεται και να χρησιμοποιείται. Τελευταίο στοιχείο τώρα. Όταν το ΝΑΤΟ προτίθεται να αναμειχθεί σε πολιτικές ε, δυνατότητες, σε πολιτικό σχεδιασμό και δράσεις, με το στρατιωτικό πολιτικό ε, προγραμματισμό είχαμε τον ενιαίο υπεύθυνο, ας το πω έτσι, ξεχωριστά υπεύθυνο. Δεν χρειάζεται αν έχουμε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικό σχεδιασμό να αναμειγνύεται το ΝΑΤΟ. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και αντίστροφα φυσικά. Μην αναμειγνιόμαστε εμεί στο ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ. Ε, ε, merci, Monsieur Gualtieri. Ευχαριστώ. Και εγώ κρίνω πάρα πολύ θετικά την έκθεση αυτή, την πάρα πολύ πλούσια, με επιχειρήματα τα οποία ε, έλκουν, αν θέλετε, τη βαθική προβληματική των περισσότερων. Συμφωνώ ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στη θεματική, γιατί διαφορετικά ο πειρασμός να επεκταθούμε ε, στα, σε ένα τόσο ζωτικό θέμα, στα πλαίσια της ΚΕΠΑ, είναι πολύ μεγάλος να ξεφύγουμε δηλαδή το συγκεκριμένο θέμα των, ε, της έκθεσης που αφορά τις πολιτικο-στρατιωτικές συνεργασίες και θεωρώ πολύ σωστό ότι κρατηθήκαμε σε αυτό το επίπεδο σε ό,τι αφορά δηλαδή και αυτή τη ρήτρα ε, είναι πολύ σημαντικό όπως είπε ο συνάδελφος Γκάλερ ίσως όμως θα ήταν καλύτερο πραγματικά να κρατήσουμε την εστίαση σε αυτή τη συγκεκριμένη πτυχή Τώρα, ερχόμαστε στα διάφορα σημεία της έκθεσης θεωρώ ζωτική σημασία το πρώτο κεφάλαιο, εκεί που μιλάμε για την θεσμική συνοχή, με αυτή την ε, σφαιρική προσέγγιση και την έμφαση που δίνεται στην ευρωπαϊκή μέθοδο αντιμετώπισης των κρίσεων στη σχέση μεταξύ της ε, πολιτικών και στρατιωτικών διαστάσεων, που ακριβώς συνεπάγεται ε, ενσωμάτωση και ενοποίηση των δύο αυτών διαστάσεων και όχι η στρατικοποίηση της πολιτικής διάστασης. Εξού και πολύ θεμητή ανησυχία την οποία εκφράζει η έκθεση ότι ίσως σε κάποια σημεία θα πρέπει ίσως να ενδυναμωθεί αυτή η εξειδίκευση, αν θέλετε, και η διατύπωση. Επί σε ό,τι αφορά τη στρατηγική πτυχή, όπου υπάρχει δηλαδή, έχει διαμορφωθεί μια τέτοια σχέση μέσω μιας δομής, της ε, δομής διεύθυνσης διαχείρισης κρίσεων και σχεδιασμού, ίσως θα μπορούσαμε περαιτέρω να ενισχύσουμε την παράγραφο που αναφέρεται στα πλαίσια των συμφωνιών που έχουν υπάρξει, η μη συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, στην χρήση εμπειριών διαχείρισης κρίσεων που προέρχονται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως είναι μέσω του μηχανισμού σταθερότητας. Να το ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το κομμάτι αυτό, γιατί ακριβώς γίνεται συζήτηση στις μέρες μας, αν είναι επαρκέ, επαρκής οι πόροι που μεταφέρονται από την Επιτροπή στην υπηρεσία που διαχειρίζεται τα θέματα βραχυπρόθεσμης σταθερότητας ή θα, μήπως θα ήταν πρόσφορο για να μην διαλύεται και διασπείρεται αυτή η τεχνογνωσία ε, που δημιουργείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχει μια δομή, ε, αν θέλετε, και μεταφορά προσωπικού σε εξωτερικό φορέα. Σε ό,τι αφορά το Γενικό Επιτελείο, συμφωνώ τη δημιουργία αυτού του επιτελείου, σχεδιασμού και εκτέλεση πολιτικών δράσεων. Εκεί όμως που γίνεται λόγος για ενοποίηση ε, λειτουργιών μεταξύ ΚΕΠΑ, στην ΚΕΠΑ μεταξύ πολιτικών και εξωτερικών δράσεων, Ίσως αυτό να προκαλεί κάποια αμφιβολία και να προκαλεί μπέρδεμα. Θα πρέπει όμως να αποσαφινιστεί ακριβώς αυτό που λέει η έκθεση, ότι δηλαδή πρόκειται ταυτόχρονα και για αξιο... να έχουμε αυτές τις δύο διαστάσεις, κεντρικές διαστάσεις, πολιτικές και εξωτικές δράσεις, δηλαδή σε επιχειρησιακό επίπεδο, που θα μπορούν να να λειτουργήσουν ταυτόχρονα, αλλά και κάθε μία να κρατά, αν θέλετε, τις που θα πρέπει να διασωθεί και να ε, διατηρείται. Δεν ξέρω εάν η υποκατάσταση αυτού του επιταλίου, του επιταλίου είναι ένα πρώτο ρεαλιστικό βήμα ή θα πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί αυτή, αυτή η έδρα από κοινού με αυτές που υπάρχουν και μετά να γίνει ενοποίηση. Δεν ξέρω μήπως είναι υπερβολικά φιλόδοξος αυτός ο, ο στόχος υποκατάστασης, αν θέλετε, και δημιουργίας αυτό το επιτέλειο όπως αναφέρεται. Γυρίζοντας πάλι πίσω, σε σχέση με την παράγραφο 3, ίσως η διατύπωση σε σχέση με την ε, αφιβολία που μπορεί να υπάρξει ότι σχεδόν πάντα χρειάζεται ταυτόχρονα πολιτική και στρατική προσέγγιση στις μεγάλες κρίσεις είναι πολύ σημαντική η συντονισμένη αυτή η προσέγγιση και είναι και ένα από τα χαρτιά, αν θέλετε, του ΝΑΤΟ. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και κρίσεις που απαιτούν αμυγός πολιτική προσέγγιση και που θα συνεχίσουν να είναι έτσι. Αλλά νομίζω ότι εδώ είναι περισσότερο θέμα διατύπωσης και όχι περιεχομένου. Σε ό,τι αφορά τα τρία άλλα κεφάλαια, συμφωνώ με τις προτάσεις, τις βρίσκω ε, κατανοητέ και τι συμμερίζομαι, επισημαίνω στη συνάδελφο Λέζινγκ ότι ο μηχανισμό της Αθήνας είναι εκτός του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας ξεχωριστός μηχανισμός, ο οποίος χρηματοδοτείται από άμεση εισφορέ των κρατών μελών. Επομένω, δεν δείχνει ζήτημα ενίσχυση του μηχανισμού αυτού από κοινού πόρους δεν, δεν λειτουργεί εις βάρος του κοινοτικού προπολογισμού, γιατί χρηματοδοτεί μόνο πολιτικές δράσεις και το διοικητικό κόστος της θεωρητικής ε, διάστασης. Και είναι σωστό αυτό που προτάθηκε και γενικά θα μπορούσαμε να πούμε και να διευρύνουμε την έννοια των πολιτικών ομάδων κρίσης, τη αντιμετώπιση κρίσεων και ενίσχυσης. Eh, των ομάδων κρούσεως δηλαδή που θα πρέπει να ε, ενισχυθούν. Όταν ενισχύεται η κοινή διάσταση χρηματοδότησης των ε, στρατιωτικών ομάδων, των ομάδων κρούσης, τόσο πιο εύκολο είναι να ενισχυθεί η συνέργεια και σε σταδικό και σε πιεσιακό επίπεδο με, τις, ε, με την πολιτική διάσταση, με τους, πολιτικούς, με τους ε, πολιτικούς μηχανισμούς. Σε ό,τι αφορά τους κοινού μηχανισμούς, συμφωνώ με τη μέθοδο πρωτίστως. Ίσως μπορούμε να συνδυάσουμε το θέμα των αποθηκών και άλλα παραδείγματα που πέραν της σωστής μεθοδολογικής προσέγγισης θα μπορούσαμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση μιας ενίσχυσης των ικανοτήτων των κοινών ε, μηχανισμών. Και τέλος, συμμερίζομαι και την παράγραφο που αφορά στο ΝΑΤΟ, σε ό,τι αφορά την πολιτική διάσταση, όπου υπάρχει κάποια αμφιβολία αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά τον ορισμό του εγγράφου που έχει εγκριθεί από τους ειδήμονες, για την νέα στρατηγική έννοια, όπου λέγονται λίγο πολύ τα πάντα και τα αντίθετά τους. Ίσως αυτή η αναφορά στην βελτίωση της ε, δομής του μηχανισμού Βερολίνο ΣΥΝ θα πρέπει να αποσαφινιστεί. Δηλαδή, προς ποια κατεύθυνση βλέπουμε αυτή τη βελτίωση. Και, εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω ότι συμμερίζομαι ε, εν γέννη την όλη προσέγγιση και γραμμή που ακολουθεί η έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Πρωτού δώσουμε το λόγο στους δύο τελευταίους συναδέλφους, η κυρία Λέζιν και πάλι, για την αλήθεια ότι σε εσά αν θέλετε στρέφονται περισσότερο τα παγιά, οπότε σα δίνουμε το λόγο. Ναι, λυπούμε που ε, σας κάνω να αισθάνεστε αμήχανος. Δεν ήταν πρόθεσή μου. Ίσως μπορείτε να το αλλάξετε εξηγώντα μου κάτι. Ίσως δεν το κατάλαβα εγώ. Θα με ενδιαφέρε να ξέρω αν μπορείτε να αναφέρετε παραδείγματα. Σε ποια σημεία. Ακριβώς σε ποια παραδείγματα στην ΑΙΤ η συνδρομή, η βοήθεια μέσω των στρατιωτικών μπόρεσε να βοηθήσει με καλύτερο τρόπο τα πράγματα από ότι αν είχαν συμμετάσχει πολιτικές δηλαδή δυνάμεις χωρίς να είναι στρατιωτικοί. Να μου εξηγήσετε γιατί χρειάστηκαν στην ΑΕΤ να πάνε πολεμικά πλοία εκεί. Φυσικά ήταν πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Ήταν ε, πλοία που είχαν και νοσοκομεία. Ήταν μεγάλα πλοία νοσοκομεία. Σε αυτά τα νοσοκομεία όμως Κανένας από τους ε, πληγωμένους της ε, IT, της IT ε, δεν, πήγαν, δεν πήγε εκεί. Τι συνέβη, οι άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να, να ξεφύγουν από αυτή τη δυστυχία της IT, τι έκαναν τα πολεμικά πλοία, αυτούς τους ανθρώπους που ήθελαν να διαφύγουν, τους ανάγκασαν να επιστρέψουν στην IT. Και γιατί χρειάστηκαν λοιπόν στρατιωτικά πολεμικά πλοία να βοηθήσουν λέει εκεί. Ίσως δεν το κατάλαβα αυτό, ίσως μπορείτε να μου το εξηγήσετε και σε σχέση με το κόστος κιόλα. Το κόστος ε, της ε, αποστολής ε, των Ηνωμένων Εθνών στην Αϊτή αν αυτά τα κόστη τα οποία για παράδειγμα τις, ε, αν δει κανείς ε, το κόστος ε, που χρειάστηκε για να αποσοβηθούν εξεγέρσεις ή επαναστάσεις στο παρελθόν, με αυτό το κόστος το οποίο δημιουργήθηκε τώρα, πώς μπορεί κανείς να δικαιολογήσει μια τέτοια κατάσταση. Ευχαριστώ. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό δηλαδή σε σχέση με τις Αμερικανικές δυνάμεις. Όμως οι Ιταλοί είχαν μία πολύ σημαντική παρουσία και η κυρία Άστον τόνισε την ε, εργασία, το έργο μάλλον ε, των Ιταλικών στρατιωτικών δυνάμεων και από τη Γουαδελούπη και την ε, Μαρτινίκα γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις και πλοία συμμετείχαν στο όλο εγχείρημα. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να δοθεί αυτή η πρώτη βοήθεια που χρειαζόταν. Συνεπώς, Δεοδός θα μπορούσαμε να έχουμε το πολιτικό σκέλος, αλλά δεν ισχύει. Αν δεν υπάρχει ένα στρατιωτικό ελικόπτερο το οποίο θα φύγει από τη Μαρτινίκα ή από τη Γουαδελούπη για να δώσει βοήθεια και αν έρθει από τη Γαλλία, χάνει κανείς 8 ώρες τουλάχιστον. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν πολύ απλοϊκό να λέμε ότι υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για στρατιωτικούς σκοπούς και ήταν εχθρικές προς τον λαό της ΑΕΤΙΣ. Τα λίγα, οι λίγες στρατιωτικές δυνάμεις που διατέθησαν τάχθηκαν υπέρ του ανθρωπιστικού έργου και αποστολών. Βεβαίως, ως προς την αποτελεσματικότητα, αυτό είναι κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, οι μόνες διαθέσιμες δυνάμεις, είτε λυπούμαστε γι' αυτό, είτε όχι, είναι στρατιωτικές δυνάμεις. Και οι Ιταλικές και οι Γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις υπηρέτησαν το λαό με την ανθρωπιστική αυτή βοήθεια. Ο κύριος Λίζεκ. Ja bardzo krótko, żeby nie powielać się argumentów i e, tez, które już zostały przedstawione przez... Είναι επαναλάβω τα επιχειρήματα που ήδη παρουσιάστηκαν από τους συναδέλφους. Θα ήθελα να αρχίσω συγχαίροντας ε, ε, για την έξοχη αυτή η έκθεση των εισηγητή. Θέλω να επιστρέψω την προσοχή σας σε δύο μικρές λεπτομέρειες. Πολλοί παρεμβαίνοντος ήδη υπογράμμισαν ότι η συνεργασία είναι απαραίτητη Στο σημείο 5 και 40 ακριβώς τονίζεται αυτή η, αναγκαι... η αναγκαιότητα, γιατί 21 από τα 28 μέλη του ΝΑΤΟ είναι κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έπρεπε λοιπόν ίσως να προσθέσουμε ότι το ποσοστό αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο αν μιλήσουμε για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων η πλειοψηφία, η συνδεπτική είναι μέλη του ΝΑΤΟ οι Πολωνοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Βρετανοί είμαστε στην, Ευρωπαϊ... είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα ως πολίτες της Ευρώπης, ταυτόχρονα μπορούμε να οριστούμε και ως ε, μέλη του ε, κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Εξού και απαιτείται η συνέργεια. Όταν ήμουν ακόμα στο Δημοτικό, κυρία Λούζινγκ, στην πρώτη Δημοτικού υπήρχε ένα εγχειρίδιο το οποίο έδειχνε διάφορα επαγγέλματα, το γιατρό, που περιποιείται τους ανθρώπους, ε, τον χτίστη που κατασκευάζει σπίτια κλπ. Και υπήρχε και μια εικόνα, ε, μια ζωγραφιά, όπου έδειχναν μια πλημμύρα και από κάτω έγραφε «Ο στρατός βοηθά τους, ε, τους πολίτες που κινδυνεύουν στις πλημμύρες». Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι και εμείς όντως στην Πολωνία, στην Τσεχική Δημοκρατία, στην καριέρα των μεγάλων καταστροφών, των πλημμυρών, χρειάστηκε να επικαλεστεί και να ζητήσει η κυβέρνηση τι στρατιωτικέ δυνάμει, γιατί αυτέ μπορούσαν να παρέμβουν αποτελεσματικά και το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστούμε κ. Σκουμουτσάκο. Ε, δύο λόγια πρώτα απ' όλα για το θέμα τη ΑΕΤ. Νομίζω ότι μια αποστολή την, την προσδιορίζει ο χαρακτήρα, ο σκοπό και ο τρόπο που αυτή εκτελείται και όχι τα μέσα με τα οποία αυτή εκτελείται. Επομένως, έτσι η επιχείρηση στην, ε, στην ΑΕΤ ήταν απολύτως μια ε, ε, επιχείρηση με πολιτική στόχευση και, και ήταν προς του πληθυσμού της ΑΕΤ. Όσον αφορά στην έκθεση, όπως ανέφερε και ο συντονιστής της ομάδας μας, ο κύριος Γκάλερ, πραγματικά είναι μια εξαιρετικά καλή έκθεση, μια πλήρης έκθεση και συγχαίρω τον εισηγητή για την δουλειά που έχει κάνει. Μια γενική παρατήρηση ε, για την από εδώ και πέρα διαδικασία. Πιστεύω και εγώ, όπως ακούστηκε προηγουμένως, ότι δεν πρέπει να υποκύψουμε στον πειρασμό να καταστήσουμε την έκθεση αυτή που έχει συγκεκριμένο αντικείμενο και συγκεκριμένο στόχο, να την καταστήσουμε μια γενική έκθεση με γενικές αναφορές στην κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Ε, και υπό αυτήν την έννοια, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η παράγραφος 42 που αναφέρεται σε ένα ε, πολιτικό ζήτημα νομίζω ότι θα μπορούσε, χωρίς να χάσει τίποτα η έκθεση από την ουσία της, να μην έχει περιληφθεί ε, στην, ε, στην έκθεση αυτή, διότι αφορά ένα ευρύτερο θέμα ε, συνεργασιών ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, τώρα, όσον αφορά στο εισαγωγικό μέρος της έκθεσης, πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο να αναφερθεί, να γίνει μια αναφορά στις δύο νέες ε, ρυθμίσεις, στις δύο νέες ρήτρες που έχει εισαγάγει οι ε, συνθήκες της Σαβώνας, δηλαδή στη ρήτρα ε, αλληλεγγύης και στη ρήτρα αμοιβαία συνδρομής. Ε, ειδικότερα τώρα για δύο παραγράφους, η παράγραφος 12 και η παράγραφος 14. Είναι πολύ θετικό ότι υπάρχει η παράγραφος 12 που αναφέρεται στο μόνιμο κέντρο επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σχέση της παραγράφου 12 με την παράγραφο 14 που προβλέπει τις ξεχωριστές διαδικασίες αποφάσεων για στρατιωτικές ή πολιτικές επιχειρήσεις. Δεδομένου ότι προβλέπονται δύο διαφορετικές, ε, δύο διαφορετικές διοικήσεις, δύο διαφορετικοί διοικητές. Ένας για στρατιωτικές επιχειρήσεις και ένας για πολιτικές επιχειρήσεις, οι οποίοι μπορούν να δρουν μέσα στο ίδιο μόνιμο κέντρο επιχειρήσεων. Εάν όμως ο τρόπος που έχουν ε, διαμορφωθεί αυτές οι παράγραφοι δημιουργεί σε συναδέλφους κάποια απορία. Νομίζω ότι ε, στην πορεία μπορεί κάποιος με πολύ μικρή προσπάθεια να διορθώσει ε, ό,τι χρειάζεται διόρθωση παρά το γεγονός ότι είναι πολύ καθαρό για να μην υπάρχουν ούτε αυτές οι πιθανές παρανοήσεις. Τέλος κύριε Πρόεδρε κλείνω με την αναφορά στην παράγραφο 43 η οποία είναι μια παράγραφος η οποία ορθώς έχει περιληφθεί και θα πρέπει να δούμε τι ε, πού ακριβώς βρίσκεται η συζήτηση στα πλαίσια του ΝΑΤΟ για την ανάπτυξη από τη Συμμαχία ε, δυνατοτήτων για, για επιχειρήσεις μη στρατιωτικές. Πιστεύω όμως ότι παράγραφος 43, όπως είναι γραμμένη, θα μπορούσε ακόμα και να ενισχυθεί προς την κατεύθυνση που έχει ε, καταγράψει ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την συμμετοχή σε αυτή την ε, πραγματιστική έκθεση δηλαδή που μας ε, παρουσιάζει πραγματικά στοιχεία. Νομίζω ότι η Κομισιόν δεν έχει τίποτα να προσθέσει ως προς αυτά τα στοιχεία. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε συμπληρωματικό ρόλο στα πλαίσια της ΠΑ, ιδιαίτερα ως προς την έρευνα και την κατάρτιση, εκπαίδευση, όπως ε, προαναφέρθηκε. Ένα γενικότερο σχόλιο σε σχέση με τη διαχείριση κρίσεων και συμμετοχή στρατιωτικών και πολιτικών δυνάμεων, στρατιωτικοπολιτικές ικανότητες δηλαδή, θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και όταν μιλάμε για εκτενή προσέγγιση δυνάμει της ε, συνθήκης της Λισαβόνας αλλά και ε, δυνάμει της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινούμαστε πέρα από το, πλαίσιο, από το στρατιωτικό πολιτικό σκέλος. Και αν μιλάμε για εκτενή προσέγγιση, μιλάμε και για πόρους που προέρχονται και από αλλού. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία ως προς τις πολιτικές επιχειρήσεις. Με πρώτη στο σκέλος, πρωταρχικό σκέλος το πολιτικό και όχι το στρατιωτικό. Κατανοώ βεβαίως ότι πολλές φορές μιλάμε για την ΚΕΠΑ η οποία έχει τα δικά της ε, χαρακτηριστικά. Πρόκειται για μια διακυβερνητική διαδικασία σε σχέση με την ε, εκτενή διαδικασία που αφορά ε, όλους τους παλαιούς πυλώνες, οι οποίοι δεν ενυπάρχουν όλοι στη συνθήκη της Λισαβόνας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Έλερ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ζωντανή αυτή θετική συζήτηση και δεν το λέω τυπικά αυτό. Έχουμε όλο το φάσμα των στοιχείων υπό τα οποία μπορεί να εξετάσει κανείς το θέμα και το καλύψαμε αυτό το φάσμα πολύ καλά. Επιμέρους επισημάνσεις τώρα. Αφενός για την κυρία Νάιτς για παράδειγμα. Το θέμα του πολιτικού δυναμικού αναφέρατε και τι θα κάνουμε. Η έκθεση νομίζω προσπαθεί συγκεκριμένες χειροπιαστές λύσεις να προτείνει και να αναφέρει. Χωρίς όμως η λογική διαχωριστική γραμμή μεταξύ ε, σχεδιασμού και εκτέλεσης στρατιωτικού και πολιτικού σκέλους ε, να ε, υπάρχει κάποια σύγχυση. Διότι είδαμε ότι υπήρξε μια μετάθεση πεδίου και που με ε, ιδιαίτερη σημασία με την συνθήκη της Λισαβόνας ε, ε, πρέπει να ληφθεί υπόψη ή με πολύ συγκεκριμένο τρόπο υπησερχόμαστε σε λεπτομέρειες τακτικού χαρακτήρα και όμως αυτά μετατίθενται σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτά που προσπάθησα εγώ να κάνω με την έκθεσή μου είναι να αναφερθώ στην πολύ συγκεκριμένη χειροπιαστή κατάσταση πώς θα αποκρισταλωθούν τώρα οι δομές που είναι αναγκαίες. Και καλείται τώρα εδώ το Ευρωκοινοβούλιο να δράσει στην δημιουργία αυτών των δομών από πλευρά του προϋπολογισμού του να μπορέσει να αρθρώσει και εκείνο τη φωνή του και τα αιτήματά του. Αυτή είναι η καταρχήν θέση μου επ' αυτών. Γι' αυτό και στο πολιτικό δυναμικό έχουμε υποβάλει προτάσεις όσον αφορά την επιμόρφωση, την κατάρτιση, όσον αφορά διαφοροποιημένες προτάσεις και για την κάλυψη δαπανών και για τον επιμερισμό δαπανών όσον αφορά κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει μόνο, ας το πω έτσι, ε, κάποια ε, επίκριση, αλλά κάνουμε συγκεκριμένες χειροπιαστές προτάσεις και δεν υπησερχόμαστε σε λεπτομέρειες, σε βάθος στις λεπτομέρειες, γιατί αυτό θα ε, διασάλευε την την ισορροπία της έκθεσης. Όσον αφορά τα battle groups, τις ομάδες κρούσης και τα Nordic, Nordic battle groups, τις σκανδιναβικές μονάδες ε, κρούσης, πρέπει εδώ να δούμε ότι σε σχέση με το, ε, την διαφοροποίηση, σε σχέση με τις standing battle groups, τις μόνιμες ε, τους μόνιμους σχηματισμούς, να δούμε να μην χαθεί αυτή η δυνατότητα, να υπάρχει σχεδιασμός και συνέχεια από πλευράς δράσεων, ώστε να διατηρούνται αυτές οι δομές. Ένα ιδιαίτερα καλό παράδειγμα σε σχέση με battle groups που διαλύθηκαν μεταξύ και δεν έχουν αφήσει πλέον ίχνη και δεν μπορεί κανείς να τις ξαναβρει. Επίσης, σε σχέση με αυτά τα προβλήματα είμαι πρόθυμος να αποσαφηνίσω τα πράγματα. Όμως, αν ξεκινήσουμε με λεπτομέρειες ευθύ εξ αρχής, τότε θα στοχοθετήσουμε πολύ γενικά θέματα Είμαι πρόθυμος να το συμπεριλάβω αυτό το θέμα, αλλά να δούμε τώρα το γιατί τα Eurocore δεν χρησιμοποιούνται και πώς αυτά σε λεπτομέρειες θα πρέπει να, εξεταστούμε, ε, να εξεταστούν. Αυτό διευρύνει ιδιαίτερα το πρίσμα. Είμαι για το μηχανισμό Αθηνά, Ατένα, ε, Είμαι ευγνώμων για τις παρατηρήσεις ε, Γκουτιέρες και σε σχέση με τον Πολ Κλοντέλ, περιβόητο πολιτιστικό ανθρωπολόγο, είπε ότι όποιος ε, θέλει να διατηρήσει ε, τα μυστικά της ε, Ανατολής, των ανατολικών χωρών, ας αποφύγει να έρθει σε ιδιαίτερα στενή επαφή με αυτά, με αυτά τα μυστικά, το μυστήριο της Ανατολής. Και τώρα σε σχέση με αυτές τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες, συνάδελφε, κατά πόσον εδώ υπάρχει ιδεολογική ε, υπερδομή από την οποία εσείς αναφέρεστε σε αυτά. Είπαμε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν χρησιμοποιούνται αυτές οι battle groups, οι ομάδες κρούσης, είναι πολιτικού χαρακτήρα. Δεν ωφελεί τώρα σε βάθος να εξετάζουμε κάθε λεπτομέρεια για κάθε ομάδα κρούσης, για, το, για ποιον λόγο δεν χρησιμοποιήθηκαν ενώ θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί. Ας μην αυταπατώμαστε. Ένας από τους κύριους λόγους των προβλημάτων των battle groups είναι ότι δεν υπάρχει ένας λογικός, ένας εύλογος, εύλογος μηχανισμός χρηματοδότησης. Και αυτό είναι μια κύρωση, μια τιμωρία την οποία εφίστανται αυτές οι ομάδες κρούσης. Πρέπει να το επισημάνουμε αυτό άλλος μηχανισμός στον οποίο μπορούμε να αναφερθούμε και στην, Λισαβόνα, στην συνθήκη Λισαβόνας δεν έχει κατοχυρωθεί. Ο μόνος μηχανισμός λοιπόν χρηματοδότησης είναι ο μηχανισμός Αθηνά. Ατένα μηχανισμός, ο μηχανισμός Αθηνά. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε τα τεχνικά προβλήματα να λύσουμε. Είναι στην ουσία χρηματοδοτικά, χρηματοοικονομικά προβλήματα, χρηματοδότησης που πρέπει να επιληθούν. Και για την IT, κοινέ προσπάθειες που έγιναν και που ε, πολλά έχουν ε, γίνει. Δεν ε, θεωρούμε ότι ήταν ιδανική η κατάσταση στην ΑΕΤ, ούτε εξειδανικεύουμε τίποτα. Αλλά σε σχέση με τα όσα έχουν αναφερθεί, το ερώτημα είναι και πρέπει να απαντηθεί συγκεκριμένα. Δεν υπάρχουν δυνατότητες, δεν υπάρχει δυναμικό στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο επίπεδο παγκόσμιας δράσης ένα αεροδρόμιο το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει να ξαναξεκινήσει. Το μόνο η μόνη δυνατότητα είναι ένα μεγάλο αεροδρόμιο με εξωτερικές τεχνικές βοήθειες, με εξωτερική τεχνική βοήθεια να μπορέσει να λειτουργήσει. Δεν θα είμαστε σε θέση χωρίς αυτό το στρατιωτικό δυναμικό τον ΗΠΑ να ανοίγαμε, να, να οδηγούσαμε στην λειτουργία ενός τέτοιου αεροδρομίου. Μπορεί κανείς να έχει διαφορετικές απόψεις για μια τέτοια δράση, αλλά και εκεί πάλι πρέπει να πει κανείς οι τηλεπικοινωνίες στην ΑΕΤ είχαν καταρρεύσει 100% και οι πρόσθετε προσπάθειες να ξαναστηθεί κάτι τηλεπικοινωνία κάστα στα πόδια του από πλευράς ενός failing state, ενός κράτους αποτυχημένου, προερχόταν από τον στρατιωτικό τομέα και σε σχέση και με τα πολεμικά πλοία, διότι εκεί μπορούσε ο τομέας των τηλεπικοινωνιών να καλυφθεί. Είναι τεράστιες οι δαπάνες που συνεπάγονται αυτές οι δράσεις. Δεν υπάρχουν πολιτικές δομές παγκόσμια αυτή τη στιγμή για μια χώρα ε, ή για ένα οποιοδήποτε εγχείρημα τηλεπικοινωνιακό ενώ κάτι έχει καταρρεύσει ξαφνικά να ξαναδημιουργηθεί και μέσα σε ε, πολύ στενό χρονικό διάστημα να αρχίσει να λειτουργεί πάλι. Και δεν υπάρχει και κανένας ε, ε, λόγος να πει κανείς ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι στρατιωτικές υποδομές. Τώρα, Όσον αφορά το ε, πολιτικό σκέλος, να πει κανείς ότι θέλουμε να το στρατιωτικοποιήσουμε, όχι, με κανένα τρόπο. Στην έκθεση δεν έχουμε ιδεολογικές ε, θέσεις ή ιδεολειψίες. Λέμε με απόλυτη κάθετη σαφήνεια ότι είναι ξεχωριστά τα δύο σκέλη, το πολιτικό από το στρατιωτικό. Στόχος μας είναι οι πολιτικές δομές, οι πολιτικές διαρθρώσεις να ενισχυθούν, να ενδυναμωθούν, να έχουν το δικό τους σκέλος και τη δική τους αλυσίδα ιεραρχίας και εντολών. Και θέλουμε στο ίδιο ιεραρχικό επίπεδο να κινούνται αυτές οι πολιτικές δράσεις στο σχεδιασμό όπως και οι στρατιωτικές. Εδώ αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Σε κάθε σημείο τονίζουμε λοιπόν την, τον αυθύπαρτο ξεχωριστό χαρακτήρα, την ε, θα έλεγα ε, ενιαία ξεχωριστή μορφή του πολιτικού σκέλους και σχεδιασμού μόνο που μεγάλες δράσεις όπως στην ΑΕΤ και αλλού δείχνουν ότι σε εναέριες μεταφορές και σε πολλά άλλα θέματα θεματολογικά δεν έχουμε πολιτικές δομές διαρθρώσεις που να μπορούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Χωρίς τις στρατιωτικές δομές δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βασιζόμαστε και χρειαζόμαστε αυτές τις στρατιωτικές υποδομές. Και όταν ασκείτε εσείς ε, κάποιες επικρίσεις πρέπει να συμφωνήσουμε ότι χωρίς αυτές τις υποδομές δεν μπορεί να γίνει τίποτα για ένα κράτος αποτυχημένο που βρίσκεται, ας το πω έτσι, ε, ισοπεδωμένο όπως ε, η ΑΕΤ στην περίπτωση αυτή. Και θα πρέπει νυφάλια και ήρεμα να δει κανεί και να αξιολογήσει το τι έγινε από όλες τις δράσεις. Όσον αφορά το θέμα αυτό το οποίο αναφέρθηκε, φυσικά πολιτικά έχει ε, ένα επίμαχο πρόβλημα, αλλά σε σχέση με το Κυπριακό και σε σχέση με το κράτος μέλος Τουρκία, αυτό τι σημαίνει. Για κάποιες δράσεις ε, στρατιωτικά επιτελεία του ΝΑΤΟ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στρατιωτικές υποδομές. Και δεν νομίζω ότι πολιτικά θα είμαστε σε θέση σε μια περίπτωση καταστροφής ε, με εκατοντάδες χιλιάδες θύματα να εξηγήσουμε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες στρατιωτικές υποδομές ή επιτελεία όπως του ΝΑΤΟ γιατί υπάρχουν λέει προβλήματα. Ε, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το θέμα ρεαλιστικά και με τα βιώματα, την εμπειρία που έχουμε σε σχέση με την Κύπρο πρέπει να δούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ξεχωριστό ε, επιτελείο. Τώρα όσον αφορά το θέμα του γενικού επιτελείου είναι επικοδομητικό και για σας κυρία Λέζινγκ να δούμε τις ε, πραγματικότητες ε, επιτόπου, το War Room της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όποιος το είδε, όποιος το επισκέφθηκε ποτέ και όχι μόνο για λόγους ασφάλειας, αλλά είναι ένας χώρος χωρίς κανένα παράθυρο που βρίσκονται ε, στον τοίχο καλώδια και όχι μόνο για όσους παρακολουθούν ταινίες του James Bond, αλλά όποιος έχει παρακολουθήσει θέματα επιμελητίας μπορεί να σκεφτεί ότι τέτοια θέματα ε, με μια, από μια τέτοια κλίμακα, ε, μέσα από μια τέτοια μονάδα όπως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεγαλύτερα ζητήματα. Πρέπει να δούμε ποια κλίμακα έχουν, ε, ποιο, εύρος έχουν αυτά τα θέματα και πώς θα είμαστε σε θέση να είμαστε στο ύψος των περιστάσεων να αναλάβουμε δράση όπως απαιτείται. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι ε, τα θέματα τα οποία αποφασίζονται να, για τα οποία αποφασίζεται να αναλυφθεί δράση ε, με χιλιάδες ε, ε στρατιώτες να μην μπορούμε μετά να κάνουμε τίποτα επειδή έχουμε κάποιο δωμάτιο όπως αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Πρέπει να δούμε πώς οι 11.000 αυτοί στρατιώτες θα μπορούσαν να οδηγηθούν και να κατευθυνθούν από ένα σωστό επιτελείο. Δεν είναι στόχος μας να δημιουργήσουμε γραφειοκρατική επιβάρυνση, ούτε θέλουμε ιδεολογικά να επιβαρύνουμε ένα θέμα. Θέλουμε να δημιουργηθούν απλά οι προϋποθέσεις, ώστε για τους στόχους που έχουμε από κοινού διατυπώσει να είμαστε αποτελεσματικοί στην δράση και στην υλοποίηση των δράσεων. Ένα τελευταίο σημείο αφορά την παράγραφο 42 και την παρατήρηση του να αφαιθεί ε, το θέμα αυτό εκτός. Είναι απλούστερο να αφαιθεί το θέμα αυτό εκτός σε σχέση με, τη, με το ΝΑΤΟ και από την Γαλλία και άλλους υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις. Μόνο που η πραγματικότητα ποια είναι. Η πραγματικότητα δεν μας αφήνει αυτό το θέμα να το αμελήσουμε, να το αφήσουμε εκτός. Πρέπει να επικεντρωθούμε με θετικά παραδείγματα. Να πούμε, χρειάζεται μια ομάδα ελικοπτέρων, ένα πουλ ελικοπτέρων και πρέπει να δράσουμε σε να διασφαλιστεί αυτή η, να καλυφθεί αυτή η ανάγκη. Και αν δεν είμαστε σε θέση από ευρωπαϊκές υποδομές σε μεγάλη κλίμακα να διασφαλίσουμε αέριες μεταφορές, ε, κάτι πρέπει να κάνουμε διότι σε περίπτωση ανάγκης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν υποδομές του ΝΑΤΟ και δεν θα είναι πάντα ουκρανικά αεροπλάνα για στρατιωτικές μεταφορές. Θα πρέπει να δούμε αν θα υπάρχει burden sharing, ένας επιμερισμός ε, βαρών με όλες τις πολιτικές ε, συνέπειες που αυτό θα συνεπάγεται στις λειτουργικές δράσεις που θα αναλαμβάνονται. Γι' αυτό το θέμα αυτό πρέπει πολιτικά με ε, ένα καθοριστικό τρόπο να αντιμετωπιστεί. Συνοψίζω, η έκθεση κάνει την προσπάθεια να μην ε, δίνει εικονικά κάποιες προτάσεις, αλλά να αναφέρεται στην πραγματικότητα, στην πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Πώς μπορούν αυτές οι διαρθρώσεις, οι δομές ε, να δημιουργηθούν και το Ευρωκοινοβούλιο να παρέμβει με θετικό τρόπο, ώστε εκεί όπου έχουμε δικαίωμα να αρθρώσουμε λόγο εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο στα θέματα των δομών και στα θέματα του σχεδιασμού να μπορέσουμε να παρέμβουμε. Χαίρομαι για τις παρεμβάσεις και προσδοκώ να δω τις τροπολογίες και είμαι πρόθυμος να συζητήσουμε και τις λεπτομέρειες και να δημιουργήσουμε μια διαφανή διαδικασία για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας όπου κυνηγάμε κάποιον και που έχει αναλάβει την σύνταξη μιας έκθεσης. Έχει την δυνατότητα το Κοινοβούλιο για πρώτη φορά να κατέβει στην κονίστρα, στην αρένα και να πει αυτές είναι οι προτάσεις που έχουμε εμείς και θέλουμε αυτές να υλοποιηθούν. Και έχουμε το πολιτικό πρόβλημα ότι έχει φιλόδοξους στόχους στην εξωτερική δράση και στην ανθρωπιστική βοήθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει στόχους που έχει διατυπώσει αλλά υπάρχει ένα κενό, ένα χάσμα μεταξύ των στοχοθετημένων αυτών δράσεων και των δυνατοτήτων και και των υποδομών μας. Αν δεν μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το gap, αυτό το χάσμα, αυτό το κενό, δεν θα είμαστε αξιόπιστοι. Θα χάσουμε την αξιοπιστία μας. Εκείνοι που περιμένουν εμείς να τους βοηθήσουμε θα απογοητευτούν και θα πιστέψουν ότι είμαστε αναξιόπιστοι. Ευχαριστώ. Ε, merci. Ευχαριστούμε. Διευκρινίζω την ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών, επόμενη Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου και δεύτερη συζήτηση έκθεσης στις 26 Οκτωβρίου πριν από την τελική έγκριση της 28 Οκτωβρίου ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Και περνάμε τώρα εντάχει στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε τον Ιούλιο στην Γεωργία με επικεφαλής τον αντιπρόεδρό μας και εισηγητή της έκθεσης του κ. Λίζικ. Dziękuję bardzo. <clears throat> Panie Przewodniczący, ponieważ Państwo macie... Ε, διαβάσατε την έκθεση της ε, αντιπροσωπείας της ε, επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία. Θα δώσω συνοπτικά τα συμπεράσματα αυτής της αντιπροσωπείας της ε, Υποεπιτροπής ε, Ασφάλειας και Άμυνας και βέβαια θα απαντήσω και στα ερωτήματά σας, εάν έχετε. Ξεκινώ λέγοντας ότι η αποστολή διήρχησε στην πραγματικότητα δύο μέρες. Στα χαρτιά διήρχησε από τις 13 έως τις 16 αλλά ταξιδέψαμε νύχτα προς τη Γεωργία. Δουλέψαμε ουσιαστικά δύο εργάσιμες ημέρες. Και αν θέλετε, ρίξτε μια ματιά στο πρόγραμμα της επίσκεψης εκείνης. Οι δύο μέρες ήταν πάρα πολύ φορτωμένες, με 7-8 συναντήσεις ημερησίως. Και θα πρέπει να, να προσθέσουμε και τις μετακινήσεις γιατί επισκεφθήκαμε τοποθεσίες όπου εργάζονται μέλη της Επιτροπής ε, Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επισκεφθήκαμε και τα λεγόμενα σύνορα. Για την ακρίβεια μια γραμμή η οποία εκτελεί χρέη συνόρου μετά την σύγκρουση και που σήμερα χωρίζει την Νότια Οσετία από την υπόλοιπη Γεωργία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εκείνης, ως αντιπροσωπεία, είχαμε τρία μέλη που εκπροσωπούσαν τα τρεις, τρεις διαφορετικές πολιτικές ομάδες, τον κύριο Παλέτσκι, τον κύριο Κόβαλ και τον υποφαινόμενο, καθώς και τον εκπρόσωπο της γραμματείας της υποεπιτροπής. Συναντήσαμε επίσης την ε, διεύθυνση της ε, αποστολής ε, παρατηρητηρίου με προσώπους του Εθνικού Κοινοβουλίου και της Κυβέρνησης της ε, Γεωργίας. Έχουμε μια μακρά, ένα μακρύ κατάλογο ονομάτων ηθινόντων. Συναντήσαμε τον Υπουργό Εσωτερικών, Εξωτερικών, Άμυνας, καθώς και την, ε, την κυρία Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας, που σήμερα είναι και πρόεδρος του Εθνικού Αυτού Συμβουλίου Ασφαλείας. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό και αυτό. Συναντήσαμε επίσης ε, βουλευτές και συγκεκριμένα τα μέλη της Επιτροπής ε, Εξωτερικών Υποθέσεων και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ήταν, συναπαρτιζόταν από μέλη και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα που συζητήσαμε, διαπιστώσαμε την απουσία μεγάλων αποκλήσεων και διαφωνιών μεταξύ του, των θέσεων του Προέδρου ε, Σακασβίλη και της αντιπολίτευσης. Οι αντιπρόσωποι της αντιπολίτευσης ε, είπαμε ότι ήταν επίσης παρόντες στη συνάντηση αυτή. Τώρα για να μιλήσουμε, οι συνομιλίες με τις νογιαγιανές αρχές ε, κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Θέσαμε προφανώς ερωτήματα συγκεκριμένα ποιο είναι το όραμα τους και η, άποψή τους, συγγνώμη, σε την εξέλιξη της κατάστασης στη Γεωργία μετά το 2008. Θέλαμε να μάθουμε ποια ήταν η άποψή του σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσει στην Γενέβη και ενδεχομένως την ένταξη της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ. Θέσαμε προφανώς ερωτήματα περί των σχέσεων ε, Γεωργίας και Ρωσίας, τις σχέσεις γειτονίας δηλαδή Γεωργίας με τη Ρωσία και μας ενδιαφέρουν και διάφορα ερωτήματα συμπεριλαμβανομένης και της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, αναφέρουμε συγκεκριμένα τη συμφωνία για την έκδοση βίζας και βέβαια τα θέματα της ανθρωπιστικής βοήθειας και των προσφύγων από την Νότια Σωτία. Όπως μπορείτε να δείτε στο πρόγραμμα το, στην προσωπία μας, επισκεφθήκαμε και χωριά προσφύγων και μιλήσαμε με πρόσφυγες κατηδίαν γιατί η αντιπροσωπεία είχε την πολύ μεγάλη τύχη να συναποδείτε από άτομα που μιλάνε αρκετά καλά ρωσικά. Δεν χρειάστηκε δηλαδή να περάσουμε από διερμηνία. Μπορέσαμε να έχουμε άμεση συζήτηση με τους πρόσφυγες αυτούς. Ε, μεγάλο τμήμα του χρόνου μας αφιερώθηκε στη συζήτηση με την διεύθυνση της αποστολής και με τους εργαζόμενους της αποστολής του μόνιμου παρατηρητηρίου και συνοδεία τους επισκεφθήκαμε αυτό που αποκαλείται σύνορο και συζητήσαμε με τους ανθρώπους εκείνους ε, για την καθημερινή τους δουλειά στα πλαίσια της αποστολής και μπορέσαμε να καταλάβουμε πώς είναι οργανωμένοι. Οφείλω να πω ότι εντυπωσιαστήκαμε από την πολύ καλή οργάνωση εργασίας της ε, αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Γεωργία. Οι γεωργιανοί προσκεκλημένοι μας μας επιβεβαίωσαν πλην Συγγνώμη, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την άποψή τους ότι λειτουργεί η αποστολή αυτή και είναι καλά προετοιμασμένη για να ασχοληθεί με περιφερειές όπου τώρα σήμερα είναι απαγορευμένη η προσπέλαση. Αυτό είναι αλήθεια και ένα από τα ατυχή συμπέρασματά μας, κάτι που μας απογοήτευσε. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Αποστολή Επιτήρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύεται να προσπελάσει την Νότια Οσετία και την Απχαζία. η κατάσταση κατά μήκο του συνόρου αυτού, εντό εισαγωγικών, κατά μήκο δηλαδή αυτή τη γραμμή οριαθέτηση, είναι καλύτερη από ό,τι ήταν πριν από λίγου μήνε ή πριν από περισσότερο πριν από ένα χρόνο. Αυτό είναι σίγουρο. Αναφέρομαι σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και θα έλεγα και κάποια σχετική ηρεμία που παρατηρείται κατά μήκο της διαχωριστικής αυτής γραμμής που χωρίζει τη Γεωργία από την Νότια Σετία. Δεν είμαι ο ίδιος διασώτης της στρατιωτικής παρουσίας των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή εκείνη. Οφείλω όμως να πω ότι και οι τρεις συμφωνήσαμε με την παρατήρηση αυτή και εξάλλου η κυρία Πρέσβης, Πρέσβης Έκλοντ της και της Πολωνίας, της Λιθουανίας και άλλοι διπλωμάτες ήταν της ίδιας ε, άποψης. Συμπεριλαμβανομένων και των Αμερικανών. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή ο έλεγχος αυτών των ε, εντοσαγωγικών συνόρων διασφαλίζεται από τους Ρώσους στρατιώτες και όχι από την ε, αστυνομία την μεθοριακή αστυνομία της Ουσιατίας σε παραδείγματι, η κατάσταση είναι ήσυχη. Δεν υπάρχουν ανταλλαγή προβολισμών. όλα έπαυσαν πριν από κάποιους μήνες. Και κλείνω υπογραμμίζοντας ότι δεν είμαι θερμός διασώτης της παρουσίας των Ρώσων στρατιωτών σε αυτή την περιοχή. Πλην όμως επικρατεί ησυχία με την παρουσία τους. Η αντιπροσωπεία μας, όπως είπα και προηγουμένως, εντυπωσιάστηκε από την πολύ καλή οργάνωση της αποστολής επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προσωπικό που εργάζεται εκεί είναι πάρα πολύ καλά καταρτισμένο. Υπάρχουν πάρα πολλοί που ήδη έχουν κάποια εμπειρία, που έχουν συμμετάσχει σε άλλες αποστολές, είτε ανθρωπιστικές, ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπάρχουν πάρα πολλοί στο προσωπικό της αποστολής που έχουν ένα παρελθόν πολιτικής υφής ή στρατιωτικής, πραγματικά λοιπόν τα καταφέρνουν πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Και μετά τους πρώτους μήνες ε, όπου έγιναν αισθητέ οι δυσκολίε, συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τον τεχνικό ξολοπλισμό. Σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε για καθαρή βελτίωση. Συνειδητοποιείται ότι πρόκειται για μια αποστολή επιτήρηση, δεν είναι στρατιωτική αποστολή. Παρ' όλα αυτά, για λόγους ασφαλείας, η Επιτροπή αυτή ήταν ε, εφοδιασμένη με τεθρακισμένα αυτοκίνητα κλπ. Το προσωπικό το οποίο εργάζεται εκεί ε, ήταν επίσης υπό προστασία και διαθέτει έναν εξοπλισμό που είναι σχεδόν στρατιωτικός, όπως το αλεξίσφαιρο γυλαίκο, κράνη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά ασχολούνται μόνο για την διασφάλιση Τη σωματική ακυριότητας του προσωπικού. Και σήμερα η κατάσταση, όπως είπα, φαίνεται αρκετά ίσχυη και σταθερή. Εμείς λοιπόν, αντιπρόσωποι, δεν είχαμε καθόλου την ε, ανάγκη να φέρουμε είτε κράτη είτε αλεξίσφαιρα βιλέκα τη διάρκεια της επίσκεψής μας. Και όπως ε, το υπογραμμίζουμε κάπου, γιατί πρόκειται μια, για έκθεση που εξεταχθεί από την Οπόλη Προσωπία, στη σελίδα 4 Έχετε πολύ άριθμα συμπεράσματα της αποστολής μας αυτής. Διαπιστώσαμε παρόλα αυτά λοιπόν και ανησυχητικά σημεία δυναμίας. Πρώτο ήταν η, απαγόρευση προσπέλασης στην Αμπχαζία και την Νότια Οσετία. Προστίθεται σε αυτά και η ανάγκη υποδομής, ε, μιας υποδομίας ε, διασυνοριακής, είδαμε με τα, με τα μάτια μας ένα τείχος το οποίο αρχίζει και υψώνεται μεταξύ Νότιας Αιτίας και Γεωργίας και άλλες εγκαταστάσεις που στο μέλλον μπορεί να δυσκολεύσουν πάρα πολύ την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων μεταξύ αιτίας και Γεωργίας. Είναι το κομμάτι που σήμερα είναι κατηλημένο, υποκατοχή. Ένα άλλο κομμάτι της αποστολίας μας, όπως είπα και προηγουμένως, αφοσιώθηκε στα ανθρωπιστικά ζητήματα, οτιδήποτε άπτωται της κατάστασης των προσφύγων και οφείλω να πω για άλλη μια φορά ότι, ε, για το ότι ε, είχαμε εντυπωσιαστεί από την ταχύτητά της, ταχύτητα με την οποία, το, με την οποία διασφαλίζεται ένα ελάχιστο συνθήκων, αποδεκτών συνθήκων. Έχουν κατασκευαστεί πάρα πολλά σπίτια, πολύ απλά, τα οποία όμως, όπως είπα, διασφαλίζουν αυτό το ελάχιστο διαμονής. Οι άνθρωποι δηλαδή μπορούν να βρουν στέγη πάνω από το κεφάλι τους, υπάρχουν κάτι στοιχειώδη έπιπλα, υπάρχει γκάζι και ηλεκτρισμός, είναι σπίτια δηλαδή τα οποία οργανώθηκαν και άνοιξαν στους πρόσφυγες σε χρόνο ρεκόρ και σήμερα το κύριο πρόβλημα είναι η ανεργία, η έλλειψη εργασίας για αυτούς τους ανθρώπους αυτοί οι πρόσφυγες ε, ομαδοποιούνται σε ένα είδος, αν θέλετε, μικρού καταβλισμού, σε ένα χώρο συγκριτικά μικρό. Από τη μια πλευρά λοιπόν το Γεωργιανό κράτος ήρθε πραγματικά στο ύψος των περιστάσεων. Εποφελήθηκε βέβαια από την βοήθεια που ήρθε το εξωτερικό. Υπάρχουν ε, ε και υπάρχουν ταυτόχρονα ε, εγκαταστάσεις παραπήγματα για την χορήγηση πρώτων βοηθειών. Από την άλλη όμως υπάρχουν και χιλιάδες άτομα που δεν έχουν τίποτα απολύτως να κάνουν, απόλυτα άνεργα και άεργα. Ε, συμπερασματικά λοιπόν, θα λέγαμε ότι πέραν αυτών που μόλις είπα, πιστεύω ότι το κυρίαρχο ερώτημα και ζήτημα είναι η αναγκαιότητα συνέχισης της αποστολής αυτής, η οποία είναι μοναδική η μοναδική διεθνής αποστολή που είναι παρούσα στο Γεωργιανό Έδαφο. Προφανώς τα πολιτικά μέσα τα οποία διαθέτουμε θα έπρεπε να μας δώσουν, να δίνουν δυνατότητα ή τέλο πάντων θα ήταν ευκταίο να μπορούμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου το πεδίο δράσης της αποστολής αυτής να μπορεί να διευρυνθεί. για να συμπεριλάβει και την Νότια Σαντία και την Απχαζία. Αλλά βέβαια αυτό είναι ένα εγχείρημα το οποίο πρέπει να θέσουμε στην Ευρωπαϊκή Δημοπλατεία. Διπλωματία. Αυτά δεν θέλω να μακρηγορήσω κύριε Πρόεδρε και ο ε, συνάδελφος κύριος Κόβατ είναι εδώ, οπότε αν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις είμαστε στη διάθεσή σας. Δεν ξέρω, Παβέλ, αν θες να προσθέσεις εσύ κάτι στην αφήγησή μου. Monsieur Koval, que... Κύριε Θέλετε να πείτε κάτι, να προσθέσετε κάτι. Σας ευχαριστώ για αυτή την ε, πλήρη εισήγηση, αυτό τον απολογισμό μάλλον. Είχαμε και τον επικεφαλή της αποστολής στη Γεωργία που μας επισκέφθηκε τον Ιούνιο και ήρθε σε επαφή με τις αρχές της Γεωργίας. Ήταν εξαιρετική η εργασία αυτής της αποστολής. Είναι η μόνη διεθνής αποστολή η οποία υπάρχει στη Γεωργία μετά την αναχώρηση των Ηνωμένων Εθνών είναι ύψης της σημασίας η παρουσία της και θα πρέπει να ε, συνεχίσει να δράμε με τον επαγγελματισμό που τη διακρίνει. Γνωρίζοντας τι συμβαίνει σε αυτή την επίμαχη περιφέρεια. Βεβαίως ε, θα πρέπει να εξευρεθεί μια πολιτική διπλωματική λύση, διότι ελοχεύει ένας πολύ μεγάλος ε, κίνδυνος, μια διπλή απογοήτευση από τις γεωργιανές αρχές σε σχέση με μια θητεία που είναι περιορισμένη. Αυτό αφορά και την φύση της αποστολής, η οποία δεν μπορεί να κινηθεί πέραν αυτής της γεωγραφικής περιφέρειας. Δεν υπάρχει ε, προσπελασιμότητα στην Οσετία και στην Απχαζία, όπως ξέρετε. Και υπάρχει και ένας ε, μεγάλος πολιτικός κίνδυνος ως προς αυτό το σκέλος. Υπάρχουν συνάδελφοι που θα ήθελαν το λόγο επί του θέματος. Όχι, όλα ήταν απόλυτα σαφή, να έχετε το λόγο, κύριος Γκουαλτιέρη. Μία ερώτηση μόνο. Σε σχέση με τις ανησυχίες και τις διαδικασίες υποστήριξης από ορισμένε χώρες και το γεγονός ότι θα πρέπει να δούμε ορισμένους ε, κανόνες που αφορούν την ε, ε, αποστολή αυτή και την επιβολή των κανόνων της ΕΠΑΤΗ εννοούσατε ως προς αυτό το σημείο. Πράγματι, ε, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το θέμα αφορούσε την χώρα μου, την Πολωνία και με ενόχλησε κάπως αυτό. Δηλαδή το προσωπικό ε, δεν, έχει, δεν κατέχει μια συγκεκριμένη θέση στην χώρα προέλευσης. Δηλαδή μετά από ένα χρόνο θα πρέπει να επανέλθει αυτό το προσωπικό στην Πολωνία για να μπορέσει να συνεχίσει να συμμετέχει στην αποστολή. Αλλά αυτό είναι μια εσωτερική υπόθεση, ήδη αναφέρθηκα σε αυτήν στον δικό μας ΙΠΕΞ. Είναι ένα θέμα συνέχειας, αν θέλετε, ε, συνέχειας εργασίας, της εργασίας της, ε, της επαγγελματικής δηλαδή δραστηριότητας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό προσωπικό και θα ήταν σκόπιμο να μπορούν, ε, αυτά, να μπορούν αυτά τα πρόσωπα να παραμείνουν επί τόπου πάνω από ένα χρόνο, αλλά δεν το επιτρέπει ο πολωνικός νόμος. Ε, ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Αν δεν υπάρχουν ε, άλλες παρεμβάσεις ε, για τη Γεωργία, παραμένουμε σε αυτό το σημείο. Αύριο θα βρεθούμε στις 9 το πρωί μαζί με την ΑΦΕΤ και τους εκπροσώπους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα ήθελα οι συντονιστές να παραμείνουν λίγα λεπτά. Θα γίνει μία συνεδρίαση